θα επισυναυθεί στα συνοπτικά πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και αν μέχρι την έγκρισή τους δεν υπάρξει αντίρρηση, η διαφωνία θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Αυτές οι προτάσεις δηλαδή για τους διορισμούς. Και πάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης που είναι δήλωση της Αντιπροέδρου